συζήτηση αυτή και πάμε στο επόμενο θέμα στη μέση διάταξη που είναι οι παρεμβάσει διάρκεια ενό λεπτού. Uh, first speaker uh, is uh, Mrs. πρώτη ομιλήτρια είναι η κυρία Σόιδροβα. Děkuji, vážená paní kolegyně a kolegové. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συνάδελφοι, ένα μεγάλο θέμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η μεταναστευτική κρίση, αλλά δεν βλέπω να υπάρχει μεγάλη αλλαγή σε ό,τι αφορά την προστασία των εξωτερικών συνόρων και σε ό,τι αφορά την ειρήνη στην ε, Μέση Ανατολή. Είναι πραγματικά διανόητο το γεγονός ότι ακόμα όταν έχουμε αποφασίσει για την ασφάλεια των εξωτερικών συνόρων, ενώ ψηφίστηκαν και αποφασίστηκαν τόσο γρήγορα οι ποσοστώσεις κατανομής, υποχρεωτικές. Στην Τσεχία εθελοντικά υποδεχόμαστε πρόσφυγες, ακόμα και αν είναι σε πιο μικρό αριθμό από ό,τι στη Γερμανία και σε άλλες χώρες και υποστηρίζουμε το Ίδρυμα το οποίο στην Τσεχία έχει τοποθετήσει 150 κοινού σε συγκεκριμένες οικογένειες και χαιρόμαστε που υποστηρίζουν τόσο πολύ την κατάσταση και φυσικά υπάρχουν και ε, Αντιστάσει, αλλά εν πάση περιπτώσει επιδεικνύουμε μεγάλη αλληλεγγύη. Όσο πιο μεγάλη συνέπεια λοιπόν υπάρχει στην αντιμετώπιση μα στην Ευρώπη για την αντιμετώπιση τη κρίσης, τόσο πιο μεγάλα θα είναι και αντικτυπώ ε, από τι δράσει των κρατών και των οργανισμών. Ευχαριστώ πολύ. Το Ιταλικό σύστημα ε, διαχείρισης των επιχειρήσεων γίνεται ε, στις θαλάσσιες περιοχές ε, όπου υπάρχουν ε, πολλές εταιρείες που ασχολούνται με αυτήν ε, την διαδικασία, κυρίως οικογενειακές εταιρείες και τώρα καλούνται να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις ε, της ακύρωσης του, δικαίωμας, του δικαιώματός τους επιμονής ενώπιον της δικαιοσύνης έχουν απορριφθεί έχουν απορριφθεί οι δυνατότητες υπεράσπισης τους κόντρα στις επιπτώσεις της ε, οδηγίας Μπόλκεσταν. Γνωρίζουν ότι το μέλλον της οικογένειάς τους σε σχέση με την ελεύθερη παροχή ε, ε, υπηρεσιών είναι κάτι το οποίο δεν μπορούν να ασκήσουν. Πρόκειται για ε, περιοχές ε, λεωμένων και πρόκειται για προτάσεις που είναι αντίθετες με το κοινοτικό δίκαιο και που σίγουρα θα πρέπει να υποστηριχτούν. Ευχαριστώ. Κύριος Τζαμπάτσκι. Συνάδελφοι, ε, αγανακτό. για ε, ένα λόγο, για ένα φαινόμενο το οποίο παρουσιάζεται εδώ και πολλές μήνες με στα σύνορα Βουλγαρία και Ελλάδας. Επί κάποια έτη τα σύνορα αυτά τα κλείνουν οι Έλληνες αγρότες και το αποτέλεσμα είναι ότι οι Βούλγαροι επιχειρηματίες υπόκεινται μεγάλες ζημιές και άλλα άτομα από την Αυστρία, από άλλες χώρες επίσης υποφέρουν. Και εδώ φυσικά εννοώ τους ε, οδηγού φορτηγών. Θα ήθελα να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει τι εξή δράσει. Να δραστηριοποιηθεί καταρχά, να βρει μια γρήγορη λύση, γιατί είναι μεγάλο το πρόβλημα. Πιστεύω ότι οι ευρωπαϊκέ συνθήκε θα πρέπει να τηρούνται και να εκπληρούνται, γιατί τώρα πολλέ συνθήκε. Γιατί στη παρούσα φάση υπάρχει παραβίαση πολλών συνθήκων. Υπάρχει Είτε υπάρχει μάλλον ελευθερία μετακίνηση, είτε δεν υπάρχει. Γιατί αυτό το διάμεσο δεν κανένα. Ο κύριος Ράντος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, η διασύνδεση των ε, δικτύων συγκοινωνιών και μεταφορών Ευρωπαϊκής Ένωσης Βαλκανίων θα επιτρέψει καλύτερη επικοινωνία, καλύτερη συγκοινωνία και καλύτερη ένταξη τελικά των χωρών αυτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και καλύτερες διακρατικές σχέσεις. Γι' αυτό εδώ και μήνες ζητώ μαζί με άλλους συναδέλφους δήλωση για την επέκταση ε, του δικτύου TNT στις χώρες του Δυτικών Βαλκανίων. Στις αρχές του μήνα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε αντίστοιχη απόφαση, οπότε ε, θα επιτευχθούν και όλοι οι στόχοι που προανέφερα. Καλωσορίζω την απόφαση Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τη δήλωση ε, θα συνεχίσω να την προσεχωγράφω. Κύριος Χρυσόγονος, παρακαλώ. Τις μέρες αυτές γινόμαστε μάρτυρες της παραβίασης κάθε έννοιας ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Η αυστριακή κυβέρνηση συγκάλεσε μια εξωθεσμική παρασυναγωγή με τη συμμετοχή των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, οι περισσότερες από τις οποίες δεν είναι καν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με διακηρυγμένο στόχο να ασκήσει πίεση ώστε η Ελλάδα να διασφαλίσει υποτίθεται την προστασία των εξωτερικών συνόρων της ένωσης στην προσφυγική κρίση. κανείς δεν μας λέει όμως με ποιον τρόπο μπορεί να γίνει αυτό στα λίγα μίλια θάλασσας ανάμεσα στα ελληνικά νησιά του αιγαίου και στα τουρκικά παράλια χωρίς να έχουμε μαζικούς πνιγμούς ανθρώπων οι οποίοι δεν είναι εγκληματίες αλλά απλώς αναζητούν μια καλύτερη μοίρα. η πίεση δεν πρέπει να ασκηθεί προς την ελλάδα αλλά προς το καθεστώς της τουρκίας το οποίο ανέχεται τους παράνομους διακινητές παραβιάζοντας τις συμφωνίες του με την ευρωπαϊκή ένωση. πρέπει να σταματήσει η ανθελληνική ιστερία και να βρεθεί ευρωπαϊκή λύση στο ευρωπαϊκό αυτό πρόβλημα. ευχαριστώ. Thank uh, ευχαριστώ κυρία Ντάλι. Chers depuis quelques ε, ε, κυρίες και κύριοι, το τελευταίο καιρό στο επίκεντρο ε, της προσοχής μας είναι αυτό το ταμπόν που ε, επιτρέπει στις γυναίκες να έχουν καλύτερη ε, περίοδο έμεινη ρίση. Πριν από λίγο καιρό βγήκανε κάποιες μελέτες που, επιστημονικές που λένε ότι περιέχουν τοξικές και επικίνδυνες ουσίες αυτά τα είδη ε, προσωπικής υγιεινής όπως είναι τα ταμπών. Έχουν κινητοποιηθεί χιλιάδες Ευρωπαίοι ε, γυναίκες αλλά και άνδρες και ζητούν πλήρη σήμανση για το τι περιέχουν αυτά τα προϊόντα, ποια χημικά δεν αντιδρά η βιομηχανία και κρύβεται πίσω από το γεγονός ότι δεν υπάρχει ούτε εθνική ούτε κοινωνική, κοινωτική νομοθεσία που να την υποχρεώνει. Το Δεκέμβριο ρωτήθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είπε ότι δεν σκέφτεται να κάνει τίποτα. Παραμονές τη 8 η Μαρτίου που είναι η Παγκόσμια Μέρα τη γυναίκα και των Δικαιωμάτων τη, θα πρέπει να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα των καταναλωτριών, που δεν φαίνεται να είναι προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ζητώ από την Κομισιόν από τη μια να προστατεύσει τις γυναίκες και επιτέλους να έχει ε, σαφείς ε, κανόνες για να αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα. Mr. Batten. Thank you. Κύριε Μπάτεν, ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Στη συζήτηση σήμερα ακούσαμε τον κύριο Τούσκ και τον κύριο Γιούγκερ και οι δύο είπαν ότι αν οι Βρετανοί ε, υπερψηφίσουν για την ε, παραμονή του ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα μέτρα για τον κύριο Κάμερον θα πρέπει να περάσουν από νομοθεσία. Αλλά ο κύριο Τάσκ είπε ότι έλπιζε ότι θα μεταφραστούν σε νομοθεσία και θα σημαίνουν τροπολογία στην οδηγία για την ελεύθερη μετακίνηση που αποτελεί μια βασική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Κοινοβούλιο μπορεί να ψηφίσει για να αλλάξει ε, η συμφωνία. Δεν θα ξέρουμε παρά μετά το δημοψήφισμα τι θα ψηφίσει ο λαός της Μεγάλης Βρετανίας. Ο κύριος Κάμερον Λοιπόν, δεν ξέρω τι θα γίνει. Το βασικό θέμα είναι κατά πόσον ο βρετανικό λαό θέλει η χώρα του να είναι μια απλή περιφέρεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση ή αν θέλει να ξαναβρει την υπόστασή του ω ε, ένα εξαρτητό κράτο. Καλό το βρετανικό λαό να φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Τόκες. Elnök asszony, teremtés isteni rendjébe illeszkedő házasság. ευχαριστώ. Η οικογένεια και ο γάμος ε, αποτελούν πανάρχες αξίες και παραδόσεις οι οποίες ορίζονται η μη κυβερνητική οργάνωση η οποία ονομάζεται Συνασπισμό για την Οικογένεια Μανική ε, προωθεί μία διάταξη η οποία διακηρύσει ότι ο γάμος αποτελεί μία ε, απόφαση για ένωση μεταξύ ενός άνδρα και μία γυναίκας. Δεν θα πρέπει λοιπόν να επιτρέψουμε οι ελεύθερες προτιμήσεις σε ό,τι αφορά ανθρώπινα όντα και σε ό,τι αφορά την ισότητα των φύλων να υπονομεύσουν τη φυσική τάξη των πραγμάτων και την φυσική έννοια της οικογένειας. Δεκάδες χιλιάδες άτομα διαδήλωσαν και ζητώ από όλους τους συναδέλφους να υποστηρίξουν την υγιή ευρωπαϊκή κοινωνία και να προστατεύσουν το θεσμό του γάμου μεταξύ ενό άνδρα και μια γυναίκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σκόρμπετ. Uh, κύριο Σκόρμπετ, ε, η κυρία Καλησπέρα. Εγώ ήθελα να σας καταστήσω κοινωνού στο γεγονότος ότι πριν από έξι μήνες σχεδόν με μεγάλη πλειοψηφία ψηφίστηκε στο Κοινοβούλιο μια έκθεση που ζητούσε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει νομοθετική πρωτοβουλία για την αναγνώριση των γεωγραφικών προελεύσεων για μη τρόφιμα. Ε, ε αυτό έχει να κάνει με τα παραδοσιακά μας προϊόντα, ε, με θέσεις εργασίας ε, που έχουμε τεράστιο διεθνή ανταγωνισμό. Οπότε, θέλουμε, λέμε, να υποστηρίζουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η γεωγραφική ένδειξη λοιπόν είναι υπέρ και των επιχειρήσεων και των καταναλωτών που ξέρουν τι αγοράζουν, εγγυημένα πράγματα. Εδώ και χρόνια τώρα έχουμε μια μελέτη που επιβεβαιώνει, ήδη από το 2013, ε, ότι χρειάζεται, είναι σκόπιμο να έρθει μια τέτοια νομοθεσία και καλό την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιτέλους να αναλάβει τις ευθύνες της και να το κάνει, γιατί το λέει και η στρατηγική της για την εσωτερική αγορά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Thank you. Mr. Ευχαριστώ κύριε Δεμεσμάκερ. Συνάδελφοι, όποιος σιωπή συμφωνεί και όποιος σιωπή για θέματα αδικίας είναι συνυπεύθυνο. Και εμεί λοιπόν ω Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μιλάμε για του Κούρδου και την, στην Τουρκία. Χθε απογοητεύτηκα με την απάντηση τη υπατή εκπρόσωπη και του πρόσωπου του ΝΑΤΟ σε ό,τι αφορά την ερώτηση που έθεσα στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων στη Συρία. Ερντογάν ε, καταπολεμά του, ε, αυτού που καταπολεμούν το Ισλαμικό κράτο. Χθε ένα 16χρονο κορίτσι κατάφερε να ξεφύγει από τα ε, νύχια της Ισλαμικού κράτους. Ε, ο Ερντογάν λοιπόν μομαρτίζει ε, τέτοια χωριά. Δεν πρέπει να υπάρχει διάκριση μεταξύ άνδρων και γυναικών, γυναικών και παιδιών. Οι άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους και ο πόλεμος ε, του τουρκικού λαού, της τουρκικής κυβέρνησης κατά του ίδιου του λαού είναι πραγματικά ξεδιάντροπος, αλλά δεν εγκαλούμε στην τάξη των Ερντογάν. Αν λοιπόν συνεχίσουμε να σιωπούμε, μάλλον αν κάποιο συνεχίζει να σιωπεί, δεν θα πρέπει να είμαστε εμεί αυτοί. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο Σαλίμοβιτ. Σας ευχαριστώ. Η σημασία της σταθεροποίησης, της, ε, της συμφωνίας μάλλον σταθεροποίησης και σύνδεση με το Κωσυφοπέδιο είναι τεράστια. Έτσι στέλνουμε ένα σημαντικό μήνυμα ότι στηρίζουμε τις ευρωπαϊκές προσδοκίες ε, αυτού του λαού και στρώνουμε το δρόμο για ένα πιο δημοκρατικό και ευημερές Κωσυφοπέδιο. Ωστόσο, καθώς είμαστε εμείς εδώ, η συμφωνία και η ευρωπαϊκή πορεία του Κωσυφοπεδίου τίθεται σε κίνδυνο. Έχουν, ε, η αντιπολίτευση έχει ρίξει δακρυγόνα στο Κοινοβούλιο και διαμαρτύρεται Υπότιτλοι AUTHORWAVE ε, κατά των ενεργειών της νόμιμα εκλεγμένης κυβέρνησης για εφαρμογή της των ε, συμφωνηθέτων υπό τη συμφωνία αυτή. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να στείλουν ένα σαφές μήνυμα ότι η ρύθμιση των σχέσεων της Κωσυφοπαίδειας με τη Σερβία και ο σεβασμός των μειονοτήτων είναι προϋπόθεση για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση του Κωσυφοπαίδειου. Η συμφωνία θα πρέπει να γίνει σεβαστή. Οποιοδήποτε και αν κυβερνά το Κωσυφοπαίδιο σέλνοντας ένα τέτοιο μήνυμα θα καταστήσουμε ότι ότι η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση του κοσυφοπεδίου είναι πιο σημαντική από τη εσωτερική ιστορική διαμάχη για εξουσία και ότι η διαδικασία ολοκλήρωση δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για λάθο στόχου. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Ο κύριος χωρίστη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Χαλιβουργία στη ε, χώρα των Βάσκων πλήττεται και χάνονται ε, ε, χίλιες θέσεις εργασίας και έρχονται να προσθεθούν και άλλες εταιρείες που πλήττουν θεμελιώδη δικαιώματα χιλιάδων πολιτών, ανδρών και γυναικών. Γιατί, διότι είναι ανάλγητες οι πολυεθνικές και για τα εδάφη και για τους ανθρώπους και ιδιαίτερα στο Σεστάο, στο εργοστάσιο, έχουν ληφθεί ε, λάθος αποφάσεις από Βρυξέλλες, Μαδρίτη ή Καστέης. Γίνεται dumping. Ε, η ενεργειακή πολιτική ε, ε, δεν είναι σωστή και έχει νύψει τα σχήρα στη κυβέρνηση γιατί πούλησε και το 10%. Ε, οι εργαζόμενοι δεν είναι ένας παράγον, παραγωγής είναι βασικό στοιχείο. Η οικονομία θα πρέπει να είναι στην υπηρεσία των πολιτών και όχι στην υπηρεσία της ελίτ του 1%. Σας ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής, ο κύριος Βίνκλερ. Uh, thank you. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί βουλευτές, στις 21 Φεβρουαρίου γιορτάσαμε την ημέρα της ε, μητρικής γλώσσας. Δυστυχώς στη Ρουμανία όμως η Βουλή των Αντιπροσώπων ουσιαστικά πέρασε ένα νομοσχέδιο που δεν θα επιτρέπει στην Ουγγρική μειονότητα να χρησιμοποιεί τη γλώσσα του, τη μητρική της γλώσσας στις ε, επίσημε διαδικασίε. Αυτό δεν συνάδει ούτε με τα θεμελιώδη δικαιώματα που προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε και με το Σύνταγμα τη Ρουμανία. Θα ήθελα λοιπόν να εκφράσω στο σημείο αυτό την επιθυμία μου να διασφαλιστεί ότι αυτό δεν θα συμβεί τελικά στη Ρουμανία. Δεν μπορεί να περάσει ένα τέτοιο νόμο σχέδιο τόσο εθνικιστικό στη φύση του, το οποίο αποκλείει μια εθνική μειονότητα. Πρόκειται για μια πρόταση η οποία θα πρέπει να καταβαρατωθεί. Η κυρία Ταντσίλα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η εφορία στη Ρουμανία ζήτησε από πέντε τηλεοπτικούς σταθμούς της ομάδας ε, Impact να ε, κενώσουν ε, την έδρα τους, να κλείσουν δηλαδή εντός πέντε εργασίμων ημερών γιατί χρωστάνε στο κράτος. Γιατί κλείνει η εφορία. Ε, τι παρεμβάσεις είναι αυτές ε, ε, κρατικές. Εμείς είμαστε όλοι ίσοι απέναντι στη δικαιοσύνη. Ε, άρχισαν να κενώνουν λοιπόν κανάλια ε, του ομίλου ΑΜΠΑΚ, η τηλεόραση ε, αντένα ένα δεν χρειάζεται, διότι αυτός ο τηλεοπτικός σταθμός νοικιάζει ε, τα γραφεία του και τα στούντιο στο συγκεκριμένο κτίριο. Λοιπόν, πέντε τηλεοπτικοί σταθμοί χρειάστηκε να κενωθούν εντό πέντε ημερών. Αυτό για μας είναι ε, απόπειρα εκφοβισμού και ε, του τύπου. Ε, μπορούμε να μιλήσουμε για διοικητικέ κυρώσεις. Πουθενά άλλου στην Ευρώπη δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Δεν μπορεί σε πέντε μέρε να μετακομίσει ολόκληρο τηλεοπτικό κανάλι. Ο κύριος Γιάκοφτσιτς. Η προσφυγική κρίση είναι κάτι το οποίο έχει εκλονίσει την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει θέσει ένα αμφιβόλο την ενότητα πάει και το Δουβλίνο, ε, απειλείται και το Σέγγεν. Ήταν τόσο ισχυρή η κρίση και τόσο σφοδρή από την αρχή ε, ε, που δεν ξέραμε πώς να αντιδράσουμε. Έρχομαι δυστυχώς να διαπιστώσω ότι ούτε σήμερα έχουμε σαφή λύση και συγκεκριμένη, γιατί δεν υπάρχει ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Δεν υπάρχει ευρωπαϊκή κοινότητα. Είναι απαράδεκτα τα πράγματα αυτά. Χώρες που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι στη Βαλκανική Οδό να ε, έχουν κάνει πολλά περισσότερα από κάποια κράτη-μέλη. Και από τα 28 κράτη-μέλη μάλιστα της πλούσιας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρειάζεται περισσότερη κοινότητα, περισσότερη αργή, Αλλιώς θα καταρρεύσει όλο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Ευχαριστώ. Η κυρία Άντερσον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 αυτή την εβδομάδα θα υποβάλω γνωμοδότηση στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ για την προστασία και βελτίωση των δικαιωμάτων των ανθρώπων με ε, αναπηρίες. Ε, θα εστιάσουμε στην πλήρη εφαρμογή της σύσταση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρία, την πλήρη εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράξης για την προσβασιμότητα, την άρση όλων των φραγμών για τους ανθρώπους με αναπηρία, την προστασία των δικαιωμάτων των πιο ευάλωτων των αναπήρων συμπεριλαμβάνοντα των αστέγων, των προσφύγων και των ετών άσυλων το, ε, η, η δήλωση της Ιρλανδίας το 1960 μας ε, υποχρεώνει να προστατεύσουμε όλους τους αδύναμους. Αυτό κάνει το Sinn Féin και ε, πιστεύω πως οι άνθρωποι με την χρειάζονται την αφοσίωσή μας και τη δέσμευσή μας και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι η αντιπροσωπεία του Sinn και η αντιπροσωπή μας στην QNGL το έχουμε όλα αυτά, το λαμβάνουμε όλα αυτά σοβαρά υπόψη. Ευχαριστώ πολύ. Uh, next speaker, Mr. Ο κύριος Πόλτσακ είναι ο επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ένα από τα πιο σοβαρά προβλήματα ε, που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη είναι χωρίς καμία αμφιβολία η τρομοκρατία. Είναι ε, Και σωστά ακούμε ότι θα πρέπει να ασχολούμαστε με τα αίτια και όχι με τις συνέπειες. Είναι απολύτως σωστό αυτό. Ποια είναι λοιπόν τα αίτια και η ρίζα. Εγώ πιστεύω ότι ένα σημαντικό παράγον είναι ακριβώς η πολιτική της Σαουδικής Αραβίας στον τομέα αυτό. Στο παρελθόν δίσταζα λίγο να τα λέω τόσο έξω από τα δόντια αυτά τα πράγματα, αλλά δεν μπορώ πια να είμαι τόσο επιφυλακτικός. Δεν χωράει καμιά αμφιβολία ότι η χώρα αυτή υποστηρίζει τρομοκρατικές ομάδες, είτε έμεσα είτε και άμεσα και μάλιστα με χρηματοδότηση. Τους τελευταίους μήνες η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, δεν μπορεί, ε, έχοντας δει όλα αυτά που έγιναν, να έθελε τυφλή και να κάνει σαν να μην τρέχει τίποτα. Ε, θα πρέπει να αλλάξει στάση η Σαουδική Αραβία και να μην υποστηρίζει τρομοκράτες είναι απειλή για μας η Σαουδική Αραβία. Ευχαριστώ. Η κυρία Σαπαρτέλ. Πρόεδρε, το δικαίωμα ε, να εκφράζει κανείς τη γνώμη του είναι αντίστοιχο με την ανεξαρτησία του τύπου και την ελευθερία. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να εξασφαλίζει την ελευθερία ε, στο περιβάλλον στο οποίο να μπορούν να ανθίσουν τα ΜΜΕ. Κάνω έκκληση στην Κομισιόν αλλά και σας συνάδελφοι πρέπει να επαγρυπνούμε και να ενεργούμε σταθερά κατά κάθε απόπειρα περιορισμού τη ελευθερία έκφραση. Θα πρέπει να ε, πούμε ποια είναι η αλήθεια να πούμε και να ενημερώνουμε το κοινό. Ωστόσο, το τελευταίο καιρό στην ε, Ρουμανία εκλήθη ε, συγκεκριμένο μέσο να εγκαταλείψει την ε, έδρα του, ε, πρόκειται για διαφωνικό σταθμό, με αποτέλεσμα να μην μπορεί πια να εκπέμπει. δεν μπορούν να παρουσιάσουν πλέον τα προγράμματά τους. Εμείς πρέπει να προστατεύσουμε την ελευθεροτυπία, όπως ορίζεται και από το άρθρο 2 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανεξάρτητος και ελεύθερος τύπος είναι απαραίτητος για την επιτυχία του ευρωπαϊκού εγχειρήματος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σπουδά. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε και κύριοι βουλευτές. Η Ευρωπαϊκή ηγεσία και οι θύνοντε από τα 27 κράτη-μέλη ε, κατέβαλαν προσπάθειες για να αποτρέψουν τον Brexit δεν ε, συμφωνώ σε ό,τι αφορά τον κοινωνικό τουρισμό, αλλά για το, τα επιδόματα τέκνων δεν μπορώ να συμφωνήσω, γιατί πρόκειται για κάτι που καθορίζονται από τη χώρα προέλευση. Τα παιδιά ήδη υποφέρουν ε, συναισθηματικά και υποφέρει και και η εκπαίδευσή τους, επειδή είναι μακριά από τους γονείς. Το επίδομα αυτό λοιπόν έρχεται στο αντιστάθμισμα. Τα Παιδιά λοιπόν τα οποία έμειναν πίσω στη Ρουμανία, οι γονείς έφυγαν και τα άφησαν πίσω για να μπορέσουν να συμβάλλουν στην οικονομία και η χώρα λοιπόν αυτή εποφελείται από τους ε, υψηλά εκπαιδευόμενους και μάλιστα εκπαιδευμένους από μηχανικούς, από γιατρούς κτλ. για τους οποίους δεν έχει δαπανίσει και τίποτα να τους εκπαιδεύσει. Και εκτός αυτού, ε, τα άτομα αυτά ε, με τι συνεισφορέ του υποστηρίζουν και την εκπαίδευση των νέων ατόμων, των νέων επιστημόνων στον Εμένο Βασίλειο. Δεν συμφωνώ λοιπόν με αυτή τη δικασία. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πανέκα, σα ευχαριστώ πολύ. Η Ευρώπη απασχολεί πάνω από 350.000 Στη Γαλλιβουργία λοιπόν και στη Σλοβακία είναι σημαντική, σημαντικός αυτός ο κλάδος. Ε, παρ' όλα αυτά λοιπόν όμως ε, οι εταιρείε αυτές ε, πρέπει να πληρούν και ψηλά πρότυπα και η Κίνα προκαλεί τεράστια προβλήματα με τις μαζικές εξαγωγές της. Και χαίρομαι που σήμερα το ΕΛΚ πρότεινε συγκεκριμένα μέτρα και απέθυνε έκκληση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ληφθούν τέτοια μέτρα. Το έχουμε δείξει και στο παρελθόν το θέμα αυτό, αλλά η κατάσταση είναι κρίσιμη και πολλές ε, καταστάσεις έχουν ε, επιδεινωθεί περαιτέρω στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως για παράδειγμα η αγορά του αλουμινίου. Τα σχετικά λοιπόν μέτρα θα πρέπει να συντονίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα πρέπει να προστατεύονται οι θέσει εργασία προκειμένου να μην χαθούν και θα πρέπει να δράσουμε γρήγορα. Ευχαριστώ κύριε Ρολά. Τον Ιούνιο οι Βρετανοί πολίτες αποφασίσουν αν θέλουν ή όχι να παραμείνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουν απολύτως τη θέση τους, αλλά όχι με κάθε τίμημα. Ε, ε, είναι πιο έφραυση η ελεύθερη κυκλοφορία και θα υπάρξει διάκριση μεταξύ Ευρωπαίων ε, πολιτών και ανησυχώ γι' αυτό. Έχω θορυβηθεί επίσης όταν μια κυβέρνηση ε, που αρνείται να υιοθετήσει το ευρώ θέλει να έχει λόγο για την ευρωζώνη. Ε, όσοι θέλουν περισσότερη ε, ολοκληρώση θα πρέπει να είναι σε θέση να προχωρήσουν. Προσοχή, να μην ανοίξουμε ε, το δρόμο σε ένα ντόμινο για να αρχίσουν και άλλες χώρες να ζητούν παρεκκλήσεις και να αποδυναμώσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να αναχθεί σε μια αγορά, σε ένα άθροισμα εθνικών εγωισμών, αλλά είναι κοινέ αξίες, ένα όραμα για αλληλεγγύη και μια ευρωπαϊκή διάσταση. Αυτό είναι η ουσία.

πάντοτε μας επιτρέπει να γιορτάζουμε τη γλώσσα μας και τον αντίκτυπο που έχει στην, στον πολιτισμό μας. Η χώρα μας θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ισότιμα όσον αφορά τη γλώσσα μας και θέλω να καλωσορίζω το ότι γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το χρησιμοποιεί ως μια ευκαιρία για να χρησιμοποιηθούν τα Ιρλανδικά. Θέλουμε όμως να επεκταθεί η χρήση των Ιρλανδικών Οι Ιρλανδοί που χρησιμοποιούν την Ιρλανδική γλώσσα, επισκέπτονται το Ευρωκοινοβούλιο και τη χρησιμοποιούν τη γλώσσα μα. Ε, ε, ποτέ δεν έχει γίνει αυτό παλιότερα. Ελπίζω πω αυτό θα έχει αντίκτυπο στι μελλοντικέ γενναίε και ότι και εκείνοι θα μπορούν και να χρησιμοποιούν την Ιρλανδική γλώσσα εδώ στο Ιρλανδικό Κοινοβούλιο. Εγώ και άλλα μέλη του Συνφέιν είμαστε αποφασισμένοι να φροντίσουμε ώστε τα Ιρλανδικά να ακούγονται περισσότερο εδώ στην Ευρώπη και στην χώρα μας. Δεν θέλουμε τα Ιρλανδικά να θεωρηθούν ως δεύτερο τη γλώσσα. Θέλουμε να είναι ισότιμοι με τα αγγλικά. Ευχαριστώ. Έτσι ολοκληρώνεται η ε, περίοδος που ήταν αφηρημένη στις μονόλεπτες παρεμβάσεις. Πρέπει να κάνω μια ανακοίνωση πριν να κλείσουμε την αποψινή σύνοδο και αυτή αφορά την ομάδα Γκουε, από την οποία έχω λάβει ένα αίτημα, ότι ο